Προχωρούμε τώρα στην εκθέξη Γκέιερ για τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2017 τμήμα 3. Κύριε Γκέγερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που τίθενται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί από τις τρέχουσες ε, συνθήκες ε, να εξαγάγει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει αυτά τα οποία υπήρχαν στην οδηγία του 2016. Με βάση την τωρινή κατάσταση θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε. Υπάρχουν οι προκλήσεις όπως ε, το προσφυγικό ζήτημα και οι οδηγίες του Συμβουλίου δεν θα μπορούν ε, να ε, αποσιωπούν αυτά τα οποία έχουν γίνει τους τελευταίους 12 ε, μήνες. Στην κατηγορία της εσωτερική και εξωτερικής πολιτικής υπάρχουν 5 εκατομμύρια ευρώ για τα θέματα των προσφύγων, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ανεπαρκή για όλους τους πρόσφυγες της Συρίας και για την υποστήριξη των κρατών μελών που υποδέχονται πρόσφυγες θα πρέπει να, να χρησιμοποιηθεί και στο σύνολό της αυτή η πίστοση. Η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί από ότι πριν από ένα χρόνο, αλλά το Συμβούλιο επανέρχεται και, προς, και προτείνει ακριβώς τα ίδια όπως και πέρυσι στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου τονίζουμε ότι δεν αρκούν τα χρήματα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ανταποκριθεί στις ανάγκες ε, των κρατών μελών. Είχε δοθεί μια αρχική πίσω στις 250 εκατομμυρίων που δεν ε, μπήκε στον προϋπολογισμό για την Τουρκία. Φέτος θα υπάρχει και άλλη μια διευκόλυνση για την Τουρκία και θα πρέπει να συνεισφέρουμε τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ. 700 εκατομμύρια ευρώ δίνονται για την ανθρωπιστική βοήθεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία σωστά λαμβάνονται. Η Τουρκία ε, δέχθηκε περισσότερους πρόσφυγες από ότι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού και είναι λογικό να συνεισφέρουμε για την ε, ε, χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων. Και η ανθρωπιστική κρίση είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε τα κράτη-μέλη μόνα τους. Όλα αυτά αποτελούν προτεραιότητες. Επομένως το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει ένα από τα δύο ή να πει ότι δεν χρηματοδοτεί πλέον κάποια από αυτές τις δράσεις ή να προσαρμόσει ε, τα μέσα τα οποία διαθέτει. Το Συμβούλιο δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε και πριν ε, δεν φτάνει το πάπλωμα για να καλύψει ε, όλες τις ανάγκες και αυτό πρέπει να το διαπιστώσουμε και να δράσουμε αναλόγως. Κάνουμε λοιπόν έκκληση προς το Συμβούλιο να λάβει υπόψη του την πραγματικότητα και να ε, λάβει τα σωστά μέτρα φέτος, όχι το 2020, φέτος για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις και τις προκλήσεις τις οποίες τώρα αντιμετωπίζουμε. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού έχει καταλήξει σε μια θετική ε, άποψη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προκλήσεις ε, που τίθενται και για την Ελλάδα με βάση ε, τα όσα της έχουν επιβληθεί από την Τρόικα και να δείξουμε αλληλεγγύη για την κρίση των προσφύγων και να έχουμε τα μέσα ευελιξίας τα οποία απαιτούνται. προτείνω να ψηφίσουμε κατά της τροπολογίας 21 ε, του ΕΛΚ αύριο. Ελπίζω και η ομάδα των Πρασίνων να μπορέσει να ψηφίσει υπέρ αυτής της έκθεσης Έχουμε μιλήσει για το πρόγραμμα ITER πολλές φορές και ξέρουμε τις ε, ανάγκες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εάν αφήσουμε κατά μέρο το πρόγραμμα ITER, θα χάσουμε πολλά από αυτά τα οποία ε, μας προσφέρει το πρόγραμμα ITER. Θα πρέπει να παρατηρούμε την εξέλιξη του προγράμματος και να δούμε κατά πόσο υπάρχουν οι δημοσιονομικές ε, προϋποθέσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες του προγράμματος εάν κάποια κονδύλια δεν τα χρησιμοποιεί το είτε, θα δούμε τι άλλες χρήσεις μπορούν να βρεθούν για αυτές τις πιστώσεις. Κύριε Γκάιερ, σας ζητούμε δύο αντιφατικά πράγματα. Πρώτον, να προσπαθήσετε να τελειώσετε την ομιλία σας και δεύτερον, να μιλάτε λιγότερο γρήγορα γιατί είναι αδύνατο να μεταφραστείτε. Καλώς. Νόμιζα ότι είχα έξι λεπτά χρόνο ομιλίας ε, και θα προσπαθήσω να ολοκλήρωσω την ε, ομιλία μου. Ψηφίστηκε η έκθεση Λαμασού το 2008 σε σχέση και με τους ε, ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η ομάδα σοφών του Μάριο Μόντι επίσης διαμόρφωσε προτάσεις. Το Συμβούλιο θα πρέπει να δείξει επικοδομητική στάση. Ξέρουμε ότι κάνει δουλειά το Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο από το να επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια, αντιγράφοντας αυτά τα οποία είχε προτείνει πέρυσι. Αυτό θα ήταν προσαρμοσμένο στις ανάγκες μιας δημοκρατικής Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία, Κύριε Γεωργίευα έχει το λόγο. Ευχαριστώ τον εισηγητή που αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο του προπολογισμού της Ένωσης για την αντιμετώπιση των κρίσεων, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να συνεχίζει να υποστηρίζει την ε, ανάκαμψη, την, ε, την ε, ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Και την, το 2017 θα είναι μια δύσκολη χρονιά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο της προσφυγικής κρίσης και της ανάγκης ένταξης των προσφύγων ενώ θα συνεχιστούν οι νέες αφήξεις, ενώ ταυτόχρονα θα χρειαστεί να υποστηρίζουμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο καλωσορίζουμε την αναγνώριση από πλευράς Κοινοβουλίου ότι η αύξηση των αναγκών και η αύξηση των πιέσεων στον προπολογισμό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο στον προπολογισμό. Τέσσερις παρατηρήσεις. Μεταναστευτική προσφυγική κρίση. Χρησιμοποιήσαμε κάθε ευελιξία, κάθε καμψία του προπολογισμού. Ευχαριστούμε γι' αυτό το Κοινοβούλιο. Αν δεν το είχατε κάνει δεν θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Όπως βλέπετε προεξοφλούμε πολλές προκλήσεις. Η τελευταία είναι η ανάγκη να υπάρξει ένα νέο εργαλείο για να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στην Ευρώπη. Θα χρηματοδοτήσουμε την διευκόλυνση για την Τουρκία. Στον προπολογισμό του 2016 ήδη έχουμε κάποιες προβλέψεις. Επενδύσαμε 95 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη επένδυση δουλεύει ήδη εκεί και έχουμε και την υποχρέωση να παράσχουμε πόρους το 2017 και το 2018. Δεύτερη παρατήρηση, μια άλλη προτεραιότητα πρέπει να ξεχνάμε, η συνέχιση της ε, εξόφλησης των ε, ε, των τιμολογιών που δεν έχουν πληρωθεί τα προηγούμενα έτη. 8 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια είναι, μειώθηκαν και θα παρουσιάσουμε την ανάλυση για την ταχύτερη μείωση των απλήρωτων λογαριασμών και τις συνέπειες για τα επόμενα έτη. Όταν γίνει η πρώτη συνάντηση του διοργανικού διαλόγου για τις πληρωμές και τις εκκρεμότητες το Μάρτιο του 2014 πριν ξεκινήσει η συζήτηση για, τον, για τις κατευθυντήρες γραμμές για τον υπολογισμό του 2017. Η τρίτη παρατήρησή μου. Αυτό που είναι σημαντικό, που έχουμε μπροστά μας και είναι σημαντικό το 2017. Πρέπει βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού ΠΔΠ να συνεχίσουμε τη, την τήρηση των ανωτάτων ορίων που, έχουν αποφασίσει, που έχει αποφασίσει η Επιτροπή βάσει τεχνικών λόγων. Θα υπάρξει ανάλυση της πρωτοβουλία για την ενέργεια των νέων και πολλές σχετικές σημαντικές πρωτοβουλίες που θα βάσει αυτή της ανάλυσης περί τα μέσα Απριλίου, σε ένα μήνα δηλαδή. Επίσης, το 2017 θα έχουμε την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε τη μείωση κατά 5% του προσωπικού. Σα ζητώ λοιπόν να τα λάβετε όλα αυτά υπόψη. Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας όπως όλοι ξέρουμε. Κλείνω τονίζοντας ότι το Κοινοβούλιο στις κατευθυντήριες γραμμές ε, ζήτησε από την Επιτροπή να ασχοληθεί με το mainstreaming του προϋπολογισμού. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το 2016 έχουμε όχι μόνο να δούμε τον υπολογισμό του 17, αλλά και την αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Δεν θα συνδέσουμε τα δύο γεγονότα αναγκαστικά, αλλά πρέπει να τα σκεφτόμαστε και τα δύο. Γιατί θα υπάρχουν επιπτώσεις του μεν προς το δε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε λοιπόν με το ΕΛΚ τον κύριο Μουρεσάν για ένα λεπτό, μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Επίτροπε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προσπάθεια την οποία έκανε, για την πρότασή του και για την καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Η έκθεση, η, οποία, η πρόταση μάλλον που έχει κατατεθεί και θα ψηφιστεί αύριο, ορίζει δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, τη συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης και δεύτερον, διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης μέσω και της μείωσης των παρανόμων μεταναστών στην Ευρώπη. Σχετικά με την οικονομική ανάκαμψη, θα υπάρξουν αρκετοί πόροι για την έρευνα, την καινοτομία, τις υποδομές, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και να οδηγηθούμε στην δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση, η θέση του Κοινοβουλίου είναι σαφής και περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές που θα υιοθετήσουμε αύριο ελπίζω με μεγάλη πλειοψηφία. Ο προϋπολογισμός είναι τμήμα της λύσης. Πρέπει να δράσει το Κοινοβούλιο και πέρυσι έδρασε γρήγορα και φέτος για την μεταναστευτική κρίση και θα πρέπει όμως και οι χώρες μέλη να, να χρηματοδοτήσουν τα ειδικά ταμεία ε, για την Αφρική, ε, για την Τουρκία κτλ. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει μια μεγάλη πλειοψηφία αύριο και να καλύψουμε τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών για τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Τόμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να συγχαρώ και εγώ τον εισηγητή να πω ότι μετά από ένα προϋπολογισμό που ψηφίσαμε με αίσθηση ευξήνης πιέζοντας τα όρια της ευελιξίας έφτασε το 17 που είναι η δοκιμασία για την θέληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει την κρίση. Έχουμε ανάγκη από απαντήσεις ε, αλληλέγγυες και δίκαιες. Τα εθνικά μέσα δεν αρκούν, πρέπει να εναρμονιστούν για να δημιουργήσουμε κοινά μέσα εκεί όπου είναι κοινέ οι δυσκολίες. Το θέμα της φύλαξης των συνόρων. Δεν μπορούμε να συντονίζουμε απλά τις δράσεις των χωρών. Χρειάζεται μια ουσιαστική κοινοτική πολιτική για τα κοινά σύνορα αν θέλουμε να διασώσουμε την ελεύθερη διακίνηση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς οικονομική προσπάθεια και τα όρια του προϋπολογισμού δεν επιτρέπουν αυτή την προσπάθεια. Να θυμίσω λοιπόν την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου ε, είναι κάτι το απαραίτητο ε, και στα πλαίσια αυτού του ανανεωμένου πλασίου θα έχουμε την δυνατότητα ανάκαμψης. Ο κύριος Άσουαρθ έχει το λόγο. Πρόεδρε, ο εισηγητής πολύ σωστά εντοπίζει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Όμως η σωστή διάγνωση δεν οδηγεί πάντοτε και σε σωστή θεραπεία. Έχω τρεις παρατηρήσεις λοιπόν. Πρώτον, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού που έχει συμφωνηθεί για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και επομένως παρά τον επίγοντα χαρακτήρα πολλών προβλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να ε, ζητάμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Η Επιτροπή έχει δίκιο που εισάγει την έννοια του προϋπολογισμού βάση απόδοσης και θα πρέπει ε, να υπάρχει η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε όσα κάνουμε. Ε, δεύτερον, κατανοώ τις ανησυχίες του εισηγητή για την ανεργία των νέων και καταλαβαίνω ότι σε εποχές κρίσης οι πολιτικοί θέλουν να δείξουν ότι ανταποκρίνονται. Εξάλλου όλοι θα ήθελαν να έχουμε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης για τους νέους. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από την εμπειρία έχουμε διδαχθεί ότι τα μέσα για την ανεργία των νέων ξεκινούν από καλές προθέσεις αλλά πολύ συχνά μας απογοητεύουν ως προς την απόδοσή τους. Αυτό το οποίο θέλουν οι νέοι και οι νέοι άνεργοι είναι μια ισχυρή δυναμική οικονομία. Και φτάνω στην τρίτη μου παρατήρηση. Καταλαβαίνω ότι δίδεται μεγάλη προσοχή στην κρίση που υπάρχει στη Γεωργία και ε, στο προσφυγικό. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανταγωνιστικότητα, η θέση εργασίας και η ανάπτυξη είναι και πρέπει να παραμείνει υπαριθμόν ένα προτεραιότητα του προπολογισμού. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά ο κύριος Ντεπχέ. Πρόεδρε, επίτροπε. Έχουμε τεράστιες προκλήσεις μπροστά μας σήμερα. Το, η πολύ μικρή ανάπτυξη, ιδίω στις επενδύσεις, με επιπτώσεις, υψηλή, υπερβολικά υψηλή ανεργία, απαράδεκτη σε επίπεδο νέων. Η μεταναστευτική ε, πίεση μετά που θέτει σε κίνδυνο την αλληλεγγύη στην Ένωση και υπονομεύει τα θεμέλια της Ένωσης. Η τρομοκρατική απειλή με τη σειρά της παραμένει μεγάλη με απειλές σφαγών και τέλος οι καταστροφές στην νότια πλευρά της Μεσογείου και την Αφρική. Ενώπιον αυτών των προκλήσεων, οι δημοσιονομικές προοπτικές για το 2017 κατά την άποψη των φιλελεύθερων είναι σαφέστατες. Πρώτον, προώθηση επενδύσεων και καινοτομία, άρα ανάπτυξη υπέρ των θέσεων εργασία. Δύο, Υποστήριξη τη ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σπονδυλική στήλη τη ευρωπαϊκή οικονομία. Τρίτον, προώθηση τη πρωτοβουλία νέων. Τέταρτον, διαχείριση και όχι απλά ε, ε, επιβίωση από την, ε, της ανθρωπιστικής της μεταναστευτικής κρίσης με ασφαλείς διαδρόμους και δίκαιη συνεργασία με τρίτες χώρες, όχι παζάρια. Πέντε. Τήρηση και σεβασμός των γεω, γεωπολιτικών εξελίξεων, των γεωπολιτικών επιλογών που προκύπτουν από, ε, την, ε, τη θέση της Υπήρου μας. Με βάση αυτές τις προτεραιότητες, ε, Πρόεδρε, θα μετάσχουμε αποφασιστικά και ενεργά στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2017. Για 1,5 λεπτά η κυρία Αγιάλα. Νεριάντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γίνεται μια διαδικασία ε, που δεν μπορεί να εκπληρωθεί κάθε χρόνο. Ενημερωνόμαστε για νέες προτεραιότητες και παράλληλα και για νέες περικοπές. Η λιτότητα πλήττει και την Επιτροπή Προϋπολογισμού όπως και τα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε επαρκείς πόρους για να εκπληρώσουμε πολιτικούς στόχους καθυστερούμε ή και ακυρώνουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητες οι επενδύσεις για την ανάπτυξη της οικονομίας και για ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίως σε εποχές κρίσης. Και έχουμε μειώσει το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο κατά 85 εκατομμύρια. Και παρότι πληττόμεθα από την ε, λιτότητα, βλέπουμε τα προτινόμενα και βλέπουμε ότι οι νέοι υποφέρουν από τις συνέπειες διότι δεν έχουμε την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Είναι υποκρισία από την πλευρά του Συμβουλίου και της Επιτροπής όταν λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν τους νέους αλλά τους κόβουν τα φτερά μειώνοντας τις πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων και από την, ε, το στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων ε, εποφελούνται οι ιδιώτες επενδυτές. Μειώνονται οι δυνατότητές μας για συνοχή. Ευχαριστώ. Κύριε Μαραγκάλη, εκ μέρους των Πρασίνων. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή έκθεση που επιβεβαιώνει το, το Κοινοβούλιο προσπαθεί να είναι, όχι ότι επιτυχάνει πάντα, μια καλύτερη εκπροσώπηση των ε, διεθνών συμφερόντων, των ε, συνολικών συμφερόντων της Ένωσης. Η έκθεση αυτή κινδυνεύει πάντα να είναι απειρχαιωμένη, διότι οι εξελίξεις τρέχουν. Θέλω να τονίσω, στόσο κάποια στοιχεία που μας βρίσκουν σύμφωνους η σύνδεση με, την, με το πι την ανάγκη αύξηση των πόρων, η καλύτερη αναφορά της χρησιμοποίησης των ίδιων πόρων και η καταβολή των απλήρωτων λογαριασμών. Εν ώψη του ορίζοντα 2000, η σύνδεση με την Ευρώπη 2020 και την Youth Employment Facility το κείμενο αυτό είναι θετικό και για το λόγο αυτό ε, μας βρίσκει σύμφωνος με μία εξαίρεση που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάννη. Ο κύριος Τζάνι, 1,5 λεπτό. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός αντιμετωπίζει δυσκολίες όπως και πάρα πολλοί ε, προϋπολογισμού χωρών της Ευρωζώνης κυρίως που υφίστανται τους περιορισμούς των Βρυξελών και την τρέλα του ενιαίου νομίσματος. Αν δεν ξεφύγουμε από αυτά δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Μια αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού είναι ουτοπική, αν και κάποια προγράμματα έχουν ανάγκη από περισσότερους πόρους. Νομίζω όμως ότι είναι λίγα τα προγράμματα στα πλαίσια των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σύμφωνα με τις θριαμβευτικές ανακοινώσεις στο σχέδιο Juncker ε, δεν είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα αλλά ε, μόνο τα ίδια τα κράτη-μέλη αποφασίζουν και επιλέγουν κάποια προγράμματα χωρίς προστιθέμενη αξία προαποφασισμένα. Οι χώρες χρησιμοποιούν πιο ελεύθερα τις επενδυτικές τους δυνατότητες χωρίς να σέβονται, ε, έτσι θα πρέπει να γίνεται, τους παράλογους ευρωπαϊκούς περιορισμούς. Ε, είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για κάποια ad hoc ε, προγράμματα όπως ε, τα εκατομμύρια που θα στείλουμε στον Ερντογάν πιστεύοντας ότι έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης. Η Ευρώπη είναι ασθενής. Ο προϋπολογισμός είναι το θερμόμετρο το οποίο δείχνει ότι πρέπει να αλλάξουν τα φάρμακα. Ζήλστρα για ένα λεπτό από την Ευρώπη των Εθνών και Ελευθεριών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αυτά τα χρήματα τα οποία δίδουμε στην Τουρκία είναι παράλογα, απαράδεκτα, όπως και στην Ελλάδα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω περισσότερο για το μέσο της ευελιξίας. Προβλέπονται ε, κάποιες πιστώσεις αλλά δυστυχώς είναι μια κακή ιδέα αυτή όταν υπάρχουν κατεπήγοντα. Πού ξέρετε αν κάτι το επίγον που συμβαίνει θα είναι το χειρότερο που θα συμβεί φέτος. Υπάρχουν πολλές φορές ε, πολλές καταστροφές σε αιτήσια βάση και έτσι τα χρήματα θα δαπανηθούν την 1η Ιανουαρίου ενώ στις 2 Ιανουαρίου το Κοινοβούλιο έλεγε ότι δεν έχουμε πια αρκετά χρήματα. Συνεπώς λοιπόν Πρόεδρε δεν μπορούμε εμείς και σε επίπεδο κρατών και σε επίπεδο ευρωπαϊκό να προβλέψουμε τις μελλοντικές κρίσεις. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει μέσω ευελιξίας. Ο κύριος Φερνάντες ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο το 1% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικός για τις επενδύσεις. Οι διοικητικές δαπάνες δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο το 6% και η προστιθέμενη συνεπώς αξία του είναι σαφής. E Ή ας σκεφτούμε τις εγγυήσεις για το επενδυτικό σχέδιο Juncker έχει ήδη φτάσει τα 50 δις και θα φτάσει στα 316. Για ορισμένες χώρες μέλη αυτό θα επιτρέψει να υπάρξουν επενδύσεις αυξημένες για πάνω από 50% και είναι κάτι το απαραίτητο για την κοινωνική συνοχή και την εδαφική συνοχή. Τα λειτουργικά λοιπόν περιφερειακά προγράμματα πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες, την ανταγωνιστικότητα και να στρέψουμε την προσοχή μας και στο ορίζοντα 2020 και άλλα προγράμματα. Υπάρχει η πρωτοβουλία για τους νέους, έχουμε και άλλα κατεπήγοντα και αναφέρομαι εδώ στην κρίση των προσφύγων. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέτημα μέσα, όλη την αλληλεγγύη, όλη την ευελιξία για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Κύριος Μάνκα. Η Ευρώπη δεν έχει τις επενδύσεις που χρειάζεται η οικονομία μας και που θα επέτρεπαν να δημιουργήσουμε απασχόληση. Γι' αυτό υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επενδύσεων που έχει στόχο επενδύσεις που δεν θα ήταν δυνατές αν δεν αναλάμβανε κάποιος ε, τον επενδυτικό κίνδυνο. Ε, οι επενδύσεις αυτές ωστόσο που χρηματοδοτούνται είναι οι, καθα... οι επενδύσεις χωρίς ε, κίνδυνο. Αυτές δεν χρειάζονται κρατική υποστήριξη, τουλάχιστον στη χώρα μου. Εμείς παρέχουμε χρηματοδότηση σε τέσσερα μη επικίνδυνα project δεν είναι δηλαδή καλή χρήση των κονδυλίων της Ένωσης το να χρηματοδοτούμε ε, ασφαλείς επενδύσεις. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πρωτοσανατολίσει κάπου αλλού τις ε, ε, επενδύσεις της. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα δημοσιονομικά μέσα που περιέχει είναι φανερό ότι δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουμε την κρίση των προσφύγων και την χαμηλή οικονομική ανάπτυξη ε, καθώς και την υψηλή ανεργία των νέων. Οι δεσμεύσει ε, για έξι δις που αναλάβαμε προς την Τουρκία και το, τα κονδύλια για τη Συρία, την Ελλάδα αλλά και ό,τι έχει να κάνει με το Horizon 2020 καθώς και την πληρωμή των καθυστερημένων θα οδηγήσουν στην ανάγκη αναθεώρησης των ε, οροφών για την περίοδο 2014-2020. Ε, Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει το ίδιο και με, πρέπει να γίνει με έναν ευρωπαϊκό φόρο ο κύριος Άρνοντ. Η έκθεση αυτή μιλάει για το πώς μπορούμε να παρακάμψουμε τους κανόνες, να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό χωρίς να παραβούμε τους κανόνες του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και τα σχετικά κατόφλια. Αυτό που θέλω να τονίσω σήμερα είναι το κομμάτι του κειμένου όπου κατηγορεί τα κράτη-μέλη για ε, ε, διπρόσωπη συμπεριφορά όταν δεν θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σοκαριστικό αυτό, διότι δεν είναι ε, ωραία αυτή η κατηγορία για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο ηγέτης είναι ο Ντέιβιτ Κάμερον. Ο Ντέιβιτ Κάμερον ο οποίος ε, αφού του έγινε Πρωθυπουργό ε, δεν ε, έχει να πει τα ίδια για τη συνθήκη της Λισαβόνας όπως πριν. Και μιλάμε για την κυβέρνηση που αλλάζει αυτά τα οποία λέει τώρα που μιλάμε για το ενδεχόμενο εξόδου της Βρετανίας από το ευρώ. δεν μπορώ να απαλλάξω ε, από τις ευθύνες της Βρετανική κυβέρνηση. Θέλουμε να βρούμε τρόπο στην έκθεση αυτή να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα ε, το 2017 και περικοπές ε, ε, ζητούνται μόνο ε, για να εξοικονομήσουμε χρήματα για άλλα κονδύλια. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να κατηγορούμε τα κράτη-μέλη για διπρόσωπη συμπεριφορά, γιατί αυτό κάνουμε και στην έκθεση, παρότι κατηγορώ τον κύριο Κάμερον ε, στη δική μου χώρα. Ευχαριστώ, κύριος Μαϊνέσκου. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι για την έκθεση αυτή. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει ε, να ξεχνάμε αυτό το οποίο θέλουμε για τον ε, προπολογισμό του 2017, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Υφίσταται πιέσει ο Ευρωπαϊκό προϋπολογισμός, ιδίω λόγω του προσφυγικού ζητήματο, και πρέπει να βρούμε λύσει ε, για να ανταποκριθούμε τι προκλήσεις τη κρίση. Δεν θα πρέπει να διακινδυνεύσουν άλλε σημαντικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, πολλά αιτήματα από την πολιτική συνοχή ε, να δοθούν κονδύλια για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό γιατί χρειαζόμαστε μια δυναμική οικονομία και ανάπτυξη για την οικονομία μας. Αν λοιπόν γίνει ανακατανομή των κονδυλίων θα δοθεί μια βραχυπρόθεσμη λύση αλλά μακροπρόθεσμα θα διακινδυνεύσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Χρειαζόμαστε δημοσιονομικούς κανόνες αποδεκτούς από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να δαπανηθούν ε, τα κονδύλια της περίοδου 2014-2020 και να μην ε, επιστραφούν από τα κράτη-μέλη. Ο προϋπολογισμός 2017 θα πρέπει και να επιφέρει τις κατάλληλες διορθώσεις στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα τα, τους ίδιους πόρους και τα αποτελέσματα του προπολογισμού βάσει ε, επιδόσεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χόφμαν. Κύριε Πρόεδρε, η βιώσιμη ανάπτυξη ε, και ε, η βιώσιμη συνεργασία για την ανάπτυξη είναι το μόνο μέσο το οποίο λειτουργεί σωστά και ε, συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της κρίσης των προσφύγων και της μετανάστευσης. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και να δοθούν τα χρήματα αυτά για την ε, ασφάλεια των συνόρων και για την ε, επιστροφή ε, προσφύγων. Εδώ ε, νομίζω ότι στρεβλώνουμε τους αρχικούς μας στόχους. Αυτά τα μέσα θα πρέπει να προέλθουν από τον προϋπολογισμό και από το ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτά τα οποία ήταν απρόβλεπτα τώρα έχουν γίνει πραγματικότητα. Και για το καταπιστευματικό Ταμείο για τη Συρία και την Αφρική πρέπει να περιμένουμε ακόμη περισσότερα από τις συνεισφορές των κρατών μελών και πρέπει να επανεξετάσουμε την κλίδα κατανομής των συνεισφορών των κρατών μελών. Κυρία Χολμάγερ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι υπάλληλοι ε, ε, των ε, θεμάτων του προϋπολογισμού που προτείνουν αυτά τα θέματα κάνουν αυτό το οποίο τους ζητούν οι κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη δεν μπορούν οι υπάλληλοι ε, τελευταία στιγμή να ε, αλλάξουν κάτι επειδή το ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να προσαρμοστούν καλύτερα στις επίγουσες ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί από τη μια εβδομάδα στην άλλη ε, να ε, έχει τεράστιες αλλαγές γιατί ε, τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να δώσουν τις αντίστοιχες οδηγίες βλέπω ε, ε, ποια είναι η τύχη του Ταμείου Μαντάτ για τη Συρία και βλέπω ότι ε, όντως για τα κράτη-μέλη υπάρχουν προβλήματα στην τήρηση του προϋπολογισμού και τα προβλήματα με τους πρόσφυγες επίσης είναι γνωστά. Ελπίζω να μπορέσετε κύριε Επίτροπε να κάνετε ένα βήμα προς τα κράτη-μέλη για να μπορέσετε να προσαρμοστείτε και στις ανάγκες των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντενανό, ένα λεπτό. Ε, τον συνάδελφο για την πρότεσή του να πω ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τα δημοσιονομικά μέσα στο ύψος των πολιτικών που θέλει να εφαρμόσει. Εμείς για το 2016 χρησιμοποίησαμε όλα τα περιθώρια Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική, γεωργική, γεωπολιτική, τρομοκρατική κρίση. Τώρα πιο ο βασιλιάς είναι γυμνός και δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τις στρατηγικές πολιτικές της Ένωσης όπως το ζωβάλι, η έρευνα, η κοινή αγροτική πολιτική κτλ. Τα δημοσιονομικά μέσα λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Τίθεται το πρόβλημα και τα κράτη πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση και την ανάγκη έβρεσης νέων πόρων. Περιμένουμε με ανυπομονησία, πολύ ανυπομονησία, τα αποτελέσματα της Επιτροπής Μόντι που θα μας επιτρέψει να οξυγονώσουμε λίγο αυτό τον προϋπολογισμό. Ο κύριος Ρούμπεκ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν για την Διεθνή Μέρα της Γυναίκας πρέπει να πούμε ότι για το 2016 ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα για τις γυναίκες στον επιχειρηματικό κόσμο και θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και για την επιχειρηματικότητα των γυναικών ε, προσφύγων και το 2017 το πρόγραμμα αυτό θα μπορέσει να ενισχυθεί και να συνεχιστεί. Ε, αυτό θα πρέπει να πούμε και προς τους αρχηγούς ε, κρατών και κυβερνήσεων όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, να μπορέσουμε να έχουμε αύξηση από το 1 στο 1,1 με 0,1% του ΑΕΠ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για την κρίση του προσφυγικού και θα μπορούσαμε να διαθέσουμε τα κονδύλια εκεί όπου η απόδοση θα είναι ε, περισσότερο ε, μεγάλη. Δεν θα πρέπει να ε, παραβλέπουμε τις ανάγκες της Τουρκίας και της Ελλάδας με τους πρόσφυγες που υποδέχεται. Ε, ζητούν κονδύλια όχι μόνο τα κρατημέρια αλλά και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να μπορούν να επιτευχθούν ε, οι καλύτερες λύσεις. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικέ λύσεις και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι πολλές εναλλακτικέ λύσεις και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώτη, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω καταρχάς τον συνάδελφο για την εξαιρετική ε, παρουσίαση που έκανε. Ε, έχω λίγο χρόνο. Καταρχάς να μιλήσω για την Τουρκία. Τέθηκε το θέμα της Τουρκίας. Όπως γνωρίζετε Επίτροπε, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών εμείς προσπαθούμε να στηρίξουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο στις αποφάσεις που καλούνται να πάρουν. Κυρία Γεωργίευα, σε εσάς ομιλώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα στην Τουρκία, όπως η ελευθερία του τύπου, ε, οι ατομικές ελευθερίες και θα πρέπει να προσπαθήσουμε με να βοηθήσουμε την Τουρκία, αλλά δεν μπορούμε να ανταγνωρίσουμε αυτά. Για το 2017 λοιπόν, όπως και το 2015 και το 2016, είναι μια χρονιά η οποία σε επίπεδο δημοσιονομικό προσπαθεί να αντιμετωπίσει κυρίως τα θέματα της μετανάστευσης. Κάνουμε τις απαραίτητες προσπάθειες, αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι το θέμα είναι κατεπήγον. Είναι ένα μόνιμο θέμα, ουσιαστικά σταθερό θέμα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Νοβακόφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πρόεδρε, επίτροπε. Κάθε χρόνο εδώ μιλάμε και θέτουμε τον προϋπολογισμό του, της Ένωσης. Παρόλο που φωνάζουν, κάνουν ρητορικοί κάποιοι συνάδελφοι, είναι καιρός τώρα να σηκώσουμε το κεφάλι μας από τα νούμερα και να δούμε τι χρειάζεται ο κόσμος. Καινοτομία, τεχνολογία, τώρα πρέπει να εντοπίσουμε ένα προϋπολογισμό που θα στηρίζεται στα αποτελέσματα και την επίδοση με αύξηση των ίδιων πόρων και με μεγαλύτερη αντοχή. Δεν είναι ώρα να λέμε ότι τα χρήματα που δαπανούμε στην ε, πρωτοβουλία των νέων είναι σπατάλη και έχω υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Ας αυξήσουμε τον προϋπολογισμό για τις επιχειρήσεις, ας αυξήσουμε την ικανότητα των κρατών μελών να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την, ε, να υποβάλουν ε, αποτελεσματικά αιτήσει για την, ε, το, 2020, το 2020. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ο προπολογισμό που ψηφίζουμε τώρα είναι το πρόσωπο που θα έχει αύριο η Ένωση. Από εμά εξαρτάται να αφήσουμε μια κληρονομιά. Ο κύριος Νεγκρέσκου. είναι σαφή αυτό το οποίο προτείνονται για τον προπολογισμό του 2017. Θέλω να προσθέσω κάτι όσον αφορά τι τροπολογίε. Είμαι μέλο τη Επιτροπή Προπολογισμών και μπορώ, δεν μπορώ να δεχθώ την επιθυμία ορισμένων συναδέλφων που αμφισβητούν την πολιτική συνοχή και τα κονδύλια τα οποία δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών τη. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στι προκλήσει της οικονομικής κρίσης και της ε, μεταναστευτικής κρίσης. Αυτό προϋποθέτει μια ενωμένη Ευρώπη, δηλαδή μια Ευρώπη με παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης, όπου και οι τοπικές κοινότητες και περιφέρειες έχουν παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης. Αυτό οδηγεί στη σταθερότητα στην Ευρώπη και ε, σταθερότητα στην Ευρώπη σημαίνει και σταθερότητα των στόχων μας μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είμαι κατά των ε, τροπολογιών που έχουν υποβληθεί και αλλά επηρεάζουν την αρχική μας πορεία. Στο πλαίσιο του Catch the Eye, Πρόεδρε, πρώτα πρώτα να τονίσω Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το 2017 θα πρέπει να επιταχυνθεί η εφαρμογή των διαφορετικών ταμείων. Το, είπα ήδη αυτό, θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσει για ένα πραγματικό επίπεδο υποχρεώσεων, επαρκές επίπεδο υποχρεώσεων, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ε, τα μη καταβληθέντα ποσά. Ο προϋπολογισμός για το 2017 είναι ένας προϋπολογισμός στον οποίο θα πρέπει να έχει περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσουμε κυρίως τα της μεταναστευτικής κρίσης. Είναι έκτακτη η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, απαιτούνται έκτακτα μέτρα, πρέπει να αυξηθούν τα όρια για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση και να βρούμε και μέτρα για να βοηθήσουμε στην υποδοχή των προσφύγων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στιγμή έχουμε σημαντικές προκλήσεις για τον προϋπολογισμό της ένωσης του. 2017. έχουμε το προσφυγικό έχουμε την ανεργία έχουμε φτώχεια και πρέπει να στηρίξουμε τις επενδύσεις για να υπάρχει ανάπτυξη. στο προσφυγικό κυρία γεωργίευα βρισκόμαστε σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40.000 εγκλωβισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Με το ρυθμό που συνεχίζει στο τέλος του μηνός θα υπάρχουν 150.000 πρόσφυγες εγκλωβισμένοι. Τα Σκόπια και η Αλβανία παράνομα έχουν κλείσει τα σύνορα. Αυτοί οι πρόσφυγες πρέπει να στηριχθούν. Η Ελλάδα είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Μέχρι στιγμής έχει δαπανίσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για το 2015 αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται επιγόντως κονδύλια για την αντιμετώπιση του προσφυγικού κονδύλια που πρέπει να πάνε και στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. δεν είναι δυνατόν να είναι κλειστά τα σύνορα και να δημιουργείται πλέον ανθρωπιστική κρίση. χρειάζονται αποφάσεις και από την κομισιόν. σας ευχαριστώ. Κύριε έχετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την συζήτηση που είχαμε σήμερα που δείχνει πόσο σοβαρό είναι το καθήκον που έχουμε μπροστά μας με πολλές πιεστικές ανάγκες στην Ευρώπη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους. Συμφωνώ λοιπόν με αυτούς που τονίζουν την ανάγκη να δώσουμε προτεραιότητα σε ανάπτυξη και να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την, την πρόκληση για την Ευρώπη. Έχουμε πραγματικά εστιάσει στα, στο να προλαμβάνουμε τα προβλήματα και γι' αυτό αλλάξουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα μεταξύ των οποίων και την ικανότητα να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο εσωτερικό τη Ευρώπη και σα το λέω ότι η Κομισιόν είχε αρχίσει να το σκέφτεται πολύ πριν αυτό εμφανιστεί σαν μια πιεστική ανάγκη για την Ελλάδα. Δεν ξέρουμε τι άλλο θα ανακύψει. Ξέρουμε ωστόσο ότι σε έναν ευάλωτο κόσμο με πιο συχνές ε, αναταραχές θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να απαντούμε με ταχύτητα, παρέχοντας ευκαιρίες να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Και κλείνω λέγοντας ότι πρώτον συμφωνώ πως ανεξάρτητα από τις πιέσεις που δέχεται ο προπολογισμό πρέπει να υπάρχει χώρος για μια ευελιξία ώστε να απαντούμε γρήγορα αν προκύπτουν ανάγκες. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτούμε με πιο δημιουργικό τρόπο το πώς θα χρησιμοποιούμε τα χρήματα. Μπορούμε να πετύχουμε περισσότερους στόχους με το ίδιο ευρώ. Με ένα παράδειγμα. Πήραμε 30 εκατομμύρια από τα 500 για να αντιμετωπίσουμε πέρσι την γαλακτοκομική κρίση για να το δώσουμε στο παγκόσμιο επισητιστικό πρόγραμμα για να αγοράσουν γάλα από μας και να το δώσουν σε πρόσφυγες. Πρέπει να σκεφτούμε πιο δημιουργικά για τον προϋπολογισμό του 2017. Τελευταία παρατήρηση. Ναι, χρειαζόμαστε χρήματα, αλλά είναι δύσκολο δύσκολο και για μας, χρειαζόμαστε περισσότερο την ενότητά μας. Όταν κοιτούμε λοιπόν τον προϋπολογισμό, δεν πρέπει να δημιουργούμε περίτες συγκρούσεις και μάχες που υπονομεύουν την ενότητα της Ένωσης που χρειαζόμαστε τόσο. Ευχαριστώ. Κύριε Γκάγια, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Μιλήσατε πάντως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που έγινε και για την υποστήριξη των συναδέλφων. Δεν έτρεψαν ερωτήσει. Ε, θα συνεχίσουμε τη δουλειά μα σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ.